Ναι. Bene, allora possiamo cominciare. Θα ξεκινήσουμε. Τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας λοιπόν, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Έχετε τη διάταξη μπροστά σας, την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, θεωρώ, θεωρείται δεκτή. Ε, ανακοινώσεις τώρα της Προέδρου. Έρχομαι στις ανακοινώσεις. Ε, αυτό που ήθελα να σας πω αφορά μια απόφαση των συντονιστών μετά από συζήτηση που είχαμε μαζί και με τη γραμματεία βέβαια, προβλέπεται η συνεδρίαση, μια συνεδρίαση έκτακτη, γιατί δεν είχαμε χρόνο στις τακτικές μας συνεδριάσεις, την Τετάρτη Οκτωβρίου από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 στις Βρυξέλλες. Εκεί θα έρθει ο Επίτροπος Έτιγκερ. Θα ενημερώσει τους συντονιστές της ΣΥΤΡΑ για τα αποτελέσματα των stress test που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Η συνεδρίαση φυσικά αυτή θα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, σε όλους τους βουλευτές. Λοιπόν, 10.30 και μισή με 12.30 και μισή, 4 Οκτωβρίου, ειδική συνεδρίαση των συντονιστών την παρουσία του Επιτρόπου Έπιγκερ για τις δοκιμασίες αντοχής. Τώρα, ξαναγυρίζω στην ημερήσια διάταξη. Η έκθεση του κυρίου Τσίτσεστερ θα ψηφιστεί σε μια άλλη συνεδρίαση, όχι σήμερα. Και περνάμε στο πρώτο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης που αφορά πάντα τον κύριο Τσίτσεστα. Απολογισμός της αντιπροσωπείας που πήγε στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τον ΕΝΙΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αντιπροσωπεία μας από τον Καλφίν και την Αμισδοτήρ και εμένα φυσικά μας συνόδευσε μέλος της γραμματείας πήγαμε στο Ηράκλειο επισκεφθήκαμε τον Ενισά τον μήνα Ιούλιο Βέβαια χάσαμε πάρα πολύ χρόνο για να πάμε και να γυρίσουμε, αλλά όντας εκεί καταφέραμε νομίζω να καλύψουμε αρκετό έδαφος. Ενημερωθήκαμε βασικά από τον Ενισά για την δραστηριότητά του. Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι στις συζητήσεις που είχαμε για τη νέα εντολή και τους όρους γύρω από τη νέα εντολή ότι είναι εύκολο να παραβλέψει κανείς την καλή δουλειά που κάνει η υπηρεσία αυτή. Μας υπενθύμησαν λοιπόν το ποιες είναι οι δραστηριότητες τους. Ε, ας μου επιτρέψετε να περάσω σε λίγες λεπτομέρειες. Ε, συμμετέχουν στην ανείχνευση των απειλών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, στην βελτίωση της αντοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιθέσεις ε, της κυβερνητικού χώρου. Έχουν επίσης ομάδες ανταπόκρισης, ε, ε, άμεσης ανταπόκρισης στον τομέα της πληροφορικής σε περιπτώσεις επιθέσεων και υπάρχει και επιπλέον δραστηριότητα την οποία αναλαμβάνουν υπέρ της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά ήταν τα οποία μας παρουσίασαν. Μας παρουσίασαν επίσης και κάποια άλλα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος θα έλεγα που έχουν σχέση με την οργανωτική της δομή, την αποστολή της, τα επιμελητιακά προβλήματα, τα προβλήματα μεταφορών, τα προβλήματα προσωπικού, πρόσληψης, συγκράτησης προσωπικού και επίσης ε, και η διαδικασία της εντολής συζητήθηκε στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει με την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της προσπάθειας την οποία κάνουμε εμείς, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια νέου τύπου εντολή πέραν αυτής της βραχυπρόθεσμης την οποία υιοθετήσαμε πέρυσι. Μετά από αυτά λοιπόν, και δεν θέλω να περάσω σε άλλες λεπτομέρειες τώρα, μπορώ να δώσω ίσως κάποιες απαντήσεις σε συναδέλφους. Είχαμε επίσης μία συνάντηση με το προσωπικό του ΕΝΙΣΑ, τους δώσαμε την δυνατότητα να θέσουν και σε μας ερωτήσεις. Πράγματι είχαν προετοιμαστεί, είχαν προετοιμάσει πολλές ερωτήσεις, προσπαθήσαμε να τις απαντήσουμε, είμαι ευγνώμων στους δύο συναδέλφους που πήραν πλήρες μέρος στη διαδικασία αυτή υπήρξε η έκφραση μιας ανησυχίας θα έλεγα για το μέλλον της υπηρεσίας αυτής, για την τοποθεσία της και το οποίο φαίνεται το μέλλον της και ποιο φαίνεται να είναι το μέλλον της γιατί και το προσωπικό συνειδητοποιεί ότι στα πλαίσια του ανανεωμένου τύπου εντολής πέρυσι αυτός λύγει το Σεπτέμβριο του 2013 και όλος ο κόσμος τελικά συγκεντρώνει την προσπάθειά του έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία έγκαιρα για τη νέα εντολή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δώσουμε τις απαντήσεις. Δεν είχαμε φυσικά απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις γιατί ε, στην παρούσα φάση διαπραγματευόμεθα με την Προεδρία επί τη βάση για της προηγούμενης προσπάθειας που έχουμε κάνει και γι' αυτό να μου επιτρέψετε μόνο να πω κάτι το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με την επίσκεψη αλλά με το θέμα περισσότερο. Είχα μια συνάντηση με την Προεδρία την προηγούμενη εβδομάδα μόλις. Συζητήσαμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν πήραμε κάποια απόφαση εμείς βέβαια. Συζητήσαμε επίσης ε, και το πιθανό χρονοδιάγραμμα για ανεπίσημου τύπου τριμερής διαλόγους και υπογραμμίσαμε επίσης κάποια από τα θέματα που εκκρεμούν και από ό,τι φαίνεται και στο Συμβούλιο τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Ακούγονται πολλές απόψεις ε, και πολλές απόψεις αποκλίνουσες μεταξύ τους. Η Κυπριακή Προεδρία θέλει να προχωρήσει με μια συγκεκριμένη εντολή μια ομάδα εργασίας και στα πλαίσια αυτής να συνεχιστούν οι συζητήσεις μαζί τους. Είχαμε επίσης και μια συνάντηση των σκιωδών την προηγούμενη Πέμπτη, όπου συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσουμε τη διαδικασία έτσι ώστε κάποια στιγμή να καταλήξουμε λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που είχαμε ξεκάθαρα ψηφίσει ήδη για το θέμα. Λοιπόν, αυτά δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω στην παρούσα φάση. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων εάν τυχόν επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ συνάδελφε δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο για το συγκεκριμένο σημείο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει συνάδελφος που θέλει να θέσει ερωτήσεις, περνάμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίτσεστερ λοιπόν για τις πληροφορίες που μας έδωσε και εξ ονόματος των υπολείπων σκιωδών που είναι απόντες. Περνάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη έκθεση την έκθεση Μπελέτ. για την ασφάλεια των δραστηριοτήτων γεώτρησης σε ανοιχτή θάλασσα. Κύριε Μπελέτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Uh, Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συνεκτικός, όσο και σαφής, αλλά και σύντομος, για να ε, υπάρξει χώρος για συζήτηση και έχουμε και τις ψηφοφορίες στις τέσσερις. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Πολλές τροπολογίες κατατέθησαν, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, στο μεταξύ, οι συνάδελφοι της Νομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν ψηφίσει τις δικές σου νομοδοτήσεις. Ξέρετε ότι είναι πάνω από γνωμοδότηση, γιατί έχουμε συναρμοδιότητες εδώ με άλλες επιτροπές. Δεν γνωμοδοτούν απλώς. Και ε, παρόλο και αν έχουμε την αποκλειστικότητα σε ορισμένα άρθρα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη Νομική. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος υποστήριξε την αλλαγή της νομικής μορφής, δηλαδή από κανονισμό σε οδηγία, που πιστεύω ότι και η δική μας Επιτροπή συμφωνεί και μάλιστα με ευρία πλειοψηφία της, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, θα δείξει αργότερα. Και στη νομική επιτροπή αξίζει να αναφερθεί και ε, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, για την, ε, τις οδηγίες για την αστική ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Στη συνέχεια, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ στα σημαντικότερα σημεία που κατατέθηκαν στις τροπολογίες. πρώτο σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοοικονομική ασφάλεια και ιδιαίτερα εδώ εννοώ την οικονομική, την τεχνική δυνατότητα ε, των εταιριών για τις δραστηριότητες ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοιχτή θαλάσσης. Πολλοί προτείνουν ε, μεγαλύτερη ευθύνη αστική ευθύνη για τις περιβαλλοντικές ε, ζημίες που θα προκληθούν να έχουν οι εταιρείε. Επίσης υπάρχουν πολλές τροπολογίες που δίνουν ιδιαίτερη προστοχή σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, ευάλωτα ας πούμε την περιοχή της Ακτικής ε, και άλλες ευαίσθητες περιοχές όπου γίνονται τέτοιες εξορίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συμβαστικές προτάσεις, Πρόεδρε, τις ερχόμενες ώρες και ημέρες. Την ε, Τετάρτη το απόγευμα συνεδριάζουν επόμενη φορά οι σκιώδησηγητές και βεβαίως με χαρά να δεχτούμε από σήμερα τις προτάσεις σας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η συμμετοχή των εργαζομένων. Όλοι μας έχουμε δεχτεί πολλές ε, παρατηρήσεις και σχόλια από τις συνδικαλιστικές ενώσεις ε, του τομέα του κλάδου αυτού που έχουν εξοργιστεί κάπως γιατί δεν ήταν ε, παρόντες στην αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλές τροπολογίες για τη συμμετοχή των εργαζομένων και πολλοί άλλοι συνάδελφοι το ίδιο. Κατατέθηκαν πολλές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι μεταξύ τους ε, αντικρουόμενες ή επίμαχε. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα γι' αυτό για τη λεγόμενη τριμερή ε, διαβούλευση με συμμετοχή και των εργαζομένων. Ε, τρίτο σημείο, ο ρόλος της ΕΜΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Και εδώ δίσταντη απόψη για το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει αυτός ο οργανισμός ή μήπως χρειάζεται νέος ευρωπαϊκός οργανισμός που θα ε, δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αρκεί η ΕΜΣΑ. Ήδη προβλέπεται στη διευρυμένη εντολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και θα το γνωρίζουν οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, μου είπαν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Μεταφορών, το ψήφισε και το Κοινοβούλιο, προβλέπεται και συμφωνήθηκε νέα εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη μα τη νέα αυτή εντολή στην έκθεσή μα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο οργανισμός αυτός σε ε, επίγουσε καταστάσει και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων. Οι συνάδελφοι της Νομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος προτείνουν να κάνει και επιθεωρήσεις ε, ο ΕΜΣΑ και να υποπτεύει και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Αυτό είναι μεγάλη διεύρυνση σημαντική της εντολής και του ρόλου του ΕΜΣΑ. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε αντίθετοι, αλλά χρειάζεται συζήτηση αυτό το θέμα και μεγαλύτερη μελέτη. γιατί από τη μία έχουμε ένα πιο φιλόδοξο ρόλο για τον ΕΜΣΑ για το πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανοιχτή θαλάσσης, αλλά από την άλλη έχουμε και το προπολογισμό. Γιατί μπορούμε να συζητήσουμε πολλά, να ψηφίσουμε, αλλά θα πρέπει και στο προπολογισμό όλα αυτά να καλύπτονται. Αλλά η Επιτροπή Προπολογισμού και ο προπολογισμό δεν ε, μα ακολουθεί στις προτάσει και ούτε έχει νόημα να φτιάξουμε ε, μια χάρτινη τίγρη που να μην έχει κανένα τίγρισμα μετά. Αυτά για τον ΕΜΣΑ. Τέταρτο. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό το. Το θέμα της επαλήθευσης από ένα τρίτο ή από μια δεύτερη αρχή. Τι σημαίνει αυτό. Ότι έχει μια μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ή φυσικού αερίου που δημιουργεί μια μικρή εταιρεία για να κάνει τη συγκεκριμένη εξόριξη που δρά αυτόνομα και ε, ξεχωριστά μέσα στον ίδιο όμιλο. Εμείς προτείνουμε να διευρυνθεί και εδώ το πεδίο για την ανεξαρτησία στην επαλήθευση. Ορισμένες ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι η ανεξάρτητη επαλήθευση είναι και όταν γίνεται από ε, δεύτερο μέρος, έτσι λέγεται, δεν χρειάζεται να είναι από τρίτο μέρος, από κάποιον ανεξάρτητο τελείως. Μπορεί να είναι εντός του ιδίου ομίλου και να θεωρείται ανεξάρτητη. Αυτό που έχει σημασία είναι η ελεγκτική αρχή ε, να είναι ξεχωριστή και αντικειμενική. Και στο συμβούλιο, ε, τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν απατώμε, ο όρος επαλήτευση από τρίτο μέρος υποχρεωτική έχει αφαιρεθεί. Δηλαδή δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάποιος τρίτος που να κάνει την επαλήτευση, αρκεί να είναι μια ανεξάρτητη ε, αρχή. Άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, τα πρότυπα για τις διεθνείς παγκόσμιες δραστηριότητες, δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 18, παράγραφος 6 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ε, είδαν πολλοί συνάδελφοι και συμφωνούν με την εκτίμηση και από διάφορες επιτροπές και από την Επιτροπή μας έχουν ε, την προσδοκία ε, ή την ελπίδα οι κοινοτικέ τουλάχιστον εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ένωση να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα και προδιαγραφέ και στι παγκόσμιε δραστηριότητε εκτό τη Ένωση. Ορισμένοι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας θέλουν να υποχρεώσουμε τις ε, ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν τέτοιες υπεράκτιες δραστηριότητες να ακολουθούν τα πρότυπά μας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μπορούμε εμεί να του αναγκάσουμε. Έχουμε κάνει την αρμοδιότητα και την εξουσία. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το θέμα. Είναι πολύ λεπτό και δεν χρειάζεται να πούμε ότι και οι αδεφερόμενοι εταιρείε του κλάδου δεν ε, έχουν ενθουσιαστεί με την πρόταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και ένα τελευταίο, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα των ορισμών. Η πρόταση για κανονισμό, εμείς ε, ίσως καταλήξουμε στην οδηγία ε, υπάρχουν θέματα ορισμών, ο φορέας εκμετάλλευσης ε, ποιος είναι, operator, πώς ορίζεται. Έχω μια παρατήρηση εδώ σύντομα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, μεγάλο ατύχημα. Πώς ορίζεται το μεγάλο ατύχημα. Ε, αν δεν απατώμε, είχαμε στα ανοιχτά ε, το Αμπερντίν, το ατύχημα Elgin αν ακολουθήσουμε τον ισχύοντα ορισμό, δεν θεωρείται μείζον ατύχημα αυτό, παρόλο που έγινε μεγάλη ζημιά και χρειάζεται ακόμα διερεύνηση. Είναι στο στάδιο ακόμα της εκπόνησης η έκθεση, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή και αυτός ο ορισμός, πώς ορίζεται το μείζον ατύχημα. Αυτά. Έχω και πολλά άλλα σχόλια να κάνω, Πρόεδρε, αλλά ας πούμε για τις αρμόδιες αρχές ή για την Αρκτική. Α, ίσως θα πρέπει να αναφέρω και το εξής. Δημοσιεύτηκε στον τύπο την περασμένη εβδομάδα αφού ψήφισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος ένα άρθρο και έλεγε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ζητά απαγόρευση, μορατόριο ε, των δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο άρθρο 3. Αλλά στην αιτιολογική σκέψη 40 η διατύπωση είναι πιο ισορροπημένη και εκεί ε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας αυτή. Και λέει, στο βαθμό που είναι εξασφαλισμένη, μάλλον που δεν είναι εξασφαλισμένη ε, η κατάλληλη αντιμετώπιση σε περίπτωση ε, ε, ατυχήματος στην Αρκτική θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μην επιτρέπουν τις εξορυκτικές δραστηριότητες ή τις ερευνητικές. Δηλαδή, από τη μια ψηφίζουμε μορατόριουμ και από την άλλη στην αιτιολογική σκέψη είναι λίγο πιο ισορροπημένη η πρόταση. Επαναλαμβάνω, εκεί έχει αρμοδιότητα αποκλειστική η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και αν δεν απατώμε... Υπάρχει και μια τροπολογία που κατατέθηκε στην Ήτρε και υποστηρίζει αυτή την άποψη για το μορατόριο για την Αρκτική. Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να συζητηθεί οπωσδήποτε. Αυτά. Σταματώ εδώ. Πρόεδρε, έλεμψη στη διάθεσή σας για τα σχόλια, τις προτάσεις και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οσκόκ, έχει στήσει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Κύριο Σκίνερ ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να είναι παρόν και τον αντικαθιστώ. Ελπίζω να μεταφέρω στους συναδέλφους τις θέσεις του σαν σκιώδης εισηγητής. Ο κύριο Σκίνερ υπογραμμίζει ότι έχει υπάρξει μια ιδιαίτερα επικοδομητική ε, σχέση με τους εκπροσώπους του εισηγητή και με τους υπόλοιπους και με την φιλελεύθερη ομάδα και με την ομάδα των συντηρητικών είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ορβηγία. Προσπαθήσαμε όμως να λάβουμε υπόψη εδώ τα συμφέροντα όλων των κρετών μελών και όχι μόνο αυτών που έχουν θαλάσσια σύνορα με ε, τα δύο αυτά κράτη και με τις χώρες που άπτονται της αρκτικής ζώνης. Ε, εκφράζει την ευαρισκιά του και ο Σκίνερ για το θέμα γύρω από το αν θα υπάρξει ε, κάποια νομοθετική ρύθμιση ή κάποια οδηγία. Ο κύριος Σκίνερ λέει ότι όλοι σχεδόν είναι ικανοποιημένοι από το κείμενο του εισηγητή το οποίο είναι κάτι που θα οδηγήσει σε μια πλήρη οδηγία και όχι τόσο σε ένα κανονισμό όπως είχε προτείνει το Συμβούλιο. Το θέμα λοιπόν αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια των τροπολογιών. Οι σοσιαλδημοκράτες λοιπόν ενδιαφέρονται και για το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων και στο συγκεκριμένο τομέα και γι' αυτό έχουμε καταθέσει ορισμένες τροπολογίες σχετικά με την συμπερίληψη ενός εκλεγμένου αντιπροσώπου για θέματα ασφαλείας. Η Βίκη Φόρντ έχει καταθέσει πάρα πολλές τροπολογίες, ορισμένες από τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε. Τις υπόλοιπες θα πρέπει να τις εξετάσουμε σε βαθύτερο επίπεδο λεπτομέρειας όσο προχωράμε στη συζήτηση. Ο κύριος Σκίνερ εδώ λέει λοιπόν ότι τελικά αυτό που έχει σημασία για την Επιτροπή μας είναι να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο έτσι ώστε να λάβει υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής μας και της Επιτροπής ε, περιβάλλοντος σχετικά με θέματα όπως θέματα ασφαλείας, ευθύνης κτλ. Ο κ. Σκίνερ θα συνεχίσει τις συναντήσεις που έχει ξεκινήσει. Θα συναντηθεί αύριο με τον Νορβηγό Υπουργό Ενέργειας και σκοπεύει να, να συναντηθεί την Τετάρτη με τους υπόλοιπους σκιώδης εισηγητές έτσι ώστε τα θέματα που μένουν σε εκκρεμότητα να τύχουν περαιτέρω συζητήσεων. Ευχαριστώ λέει η κυρία Σαρτόρη, κύριο Ζαντό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εξ ονόματος του κ. που είναι σκιώδης εισηγητής για το θέμα. Ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή γιατί δεν θα μπορέσω να ακούσω τις απαντήσεις του ή τα σχόλιά του, αλλά έχω εδώ ανθρώπους που θα το κάνουν. Λοιπόν, οδηγία ή κανονισμός. Εμείς θα μέναμε στην πρόταση της Επιτροπής, τον κανονισμό, για δύο απλούς λόγους και νομίζω ότι αυτό είχε οδηγήσει ακριβώς και την Επιτροπή στο να προτείνει τον κανονισμό. Το ότι κάποια κρατημέλη σήμερα δεν έχουν μια κάποια πολιτική και θεσμού στον τομέα της ασφάλειας στις θαλάσσιες δραστηριότητες και αυτές οι προτάσεις διευκολύνουν θα έλεγα τη λήψη μέτρων στο σύνολο των κρατών μελών με ενοποιημένο τρόπο ενώ αντίθετα θα είχαμε να διατρέξουμε τον κίνδυνο δημιουργίας διαφορετικών καταστάσεων στα διάφορα κράτη-μέλη και μια οδηγία δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί με ομοιογενή τρόπο στο σύνολο των κρατών μελών. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την πρόταση της Επιτροπής Γιούρη σχετικά με την οικονομική ευθύνη έχουν ακουστεί αρκετά ενδιαφέρουσε απόψεις και από την Επιτροπή Γιούρη και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, όπως επίσης και για τις ποινικέ κυρώσει. Το θέμα δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική ευθύνη και θα επανέλθουμε εδώ στο θέμα της Αρκτικής, αλλά και η αστική ευθύνη έχει σημασία και νομίζουμε ότι οι αδειοδοτήσεις δεν θα πρέπει να προορίζονται προς επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν τις οικονομικές εγγυήσεις που απαιτούνται έτσι ώστε να καλύψουν το δυνητικό κόστος αντιστάθμισης και καθαρισμού σε περίπτωση ατυχήματος. Για την Αρκτική. Κατανοώ αυτό το οποίο θέλει ο εισηγητής να ερμηνεύσει κατά κάποιο τρόπο την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος με κάπως πιο μετριοπαθή τρόπο. Αλλά είναι σαφές ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει εκφραστεί ξεκάθαρα για το θέμα αυτό. Και εμείς πιστεύουμε ότι η άποψη της Επιτροπής Άνβη και η άποψη ε, κάποιων κρατών μελών θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ε, στην απόφαση της Επιτροπής μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει εδώ ένας μείζον περιβαλλοντικός κίνδυνος και δεν μπορούμε εμείς να θεωρήσουμε, να εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη μας μόνο τις οικονομικές πτυχές ε, της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων στην Αρκτική. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θαλασσίας Ασφάλειας. Είναι αλήθεια ότι θα έχει να παίξει έναν σημαντικότατο ρόλο απέναντι στα κράτη-μέλη. Απαιτούνται και έχουμε ανάγκη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και επιστημονική βοήθεια στα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα συντονισμού όλων των διαδικασιών αυτών. Θα θέλαμε επίσης να έχουμε και συντονιστικές ε, δυνατότητες στην περίπτωση όπου χρειαστεί να υπάρξει μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού μετά από ατύχημα, κάτι το οποίο απευχόμεθα φυσικά. Θα συνεχίσουμε τις απαφές μας με τον εισηγητή, αλλά με κάποια στοιχεία τα οποία σας παρουσίασα και τα οποία αποκλίνουν θα έλεγα από τις απόψεις που εξέφρασε και από το πνεύμα του εισηγητή. Ευχαριστώ η Φόρντεχ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ προτιμώ οδηγία παρά κανονισμό. Θα το γνωρίζουν οι συνάδελφοι γιατί το έχουμε ξαναπεί. Και για να γίνουν υψηλότερε οι προδιαγραφές ασφαλείας και για άλλους λόγους. Για να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου. Κάποιος είπε ότι υπέβαλα πολλές τροπολογίες. Ναι, με την ιδέα να καταστεί το δυνατόν σαφέστερο το ποιο φέρει την ευθύνη για να υπάρχει δηλαδή η ασφάλεια αυτή δικαίου. Και μάλιστα και μετά την κατάθεση των τροπολογιών είχα και σχόλια από των τροπολογιών και τροπολογίες από των τροπολογιών. Άρα πράγματι ο δρόμος θα είναι μακρός. Είναι όμως πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Γνωρίζω ότι η χώρα μέλος μου έχει πολλές offshore, αλλά είναι σημαντικό και για τις ε, υπόλοιπε ε, χώρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και για τι υπόλοιπε ε, χώρε μέλη. Τώρα, για το θέμα τη Αρκτική. Είναι βέβαια ευαίσθητο το θέμα, καθώ επίση θα είναι ευαίσθητη και η διατύπωση. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τι γίνεται πιο πολύ στα ευρωπαϊκά ύδατα και να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όπου αυτό είναι δυνατό θα θέλαμε η Ευρώπη μέσω του Συμβουλίου, μέσω των χωρών μελών να απαιτήσει την εφαρμογή των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας του περιβάλλοντος και στην Αρκτική. Για την ΕΜΣΑ, για τον, η 264 τροπολογία νομίζω αποτελεί καλή βάση για την διατύπωση αυτή. Πολλοί ζητούν από την ΕΜΣΑ να κάνει διάφορα πράγματα. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί ή ότι θέλει να τα κάνει τα πράγματα αυτά. Ίσως Χρειάζεται μια συζήτηση είτε επισήμως μέσω του Προέδρου είτε και ξεχωριστά. Δεν θέλουμε να τους ε, σπρώξουμε σε κάτι που δεν θα είναι απόλυτα νόμιμο και επομένως να έχουμε ακόμα περισσότερες συζητήσεις. Ναι, να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, offshore authorities form. Γιατί δράση εκτό τη Ευρώπη φαίνεται, εκτό, Ένωση δηλαδή φαίνεται να υπάρχει γενικά υποστήριξη των τροπολογιών και για την αρχή ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια τι προδιαγραφές ασφαλεία. Εγώ έχω βαρεθεί να του ακούω να μου το λένε αυτό, έρχονται και μου το λένε διαρκώς. Χρειαζόμαστε να καταστήσουμε βέβαιο ότι με κάποιο τρόπο του ενθαρρύνουμε να τηρούν τις υψηλότερες προδιαφές ασφαλείας μεν, αλλά δεν έχουμε όμως ε, την εξουσία να τους εξαναγκάσουμε. Ούτε θέλουμε βεβαίως να τους κόψουμε τα πόδια με την έννοια να μην μπορούν να λειτουργήσουν ε, ε, υπερακτίως. Τώρα, μίλησα για την ασφάλεια δικαίου. Ίσως να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και την υπηρεσία του Κοινοβουλίου που κάνει μελέτες αντικτύπου για τα θέματα ευθύνη και Και, και να δούμε τι άλλε τροπολογίε. μένουν πολλά ερωτηματικά για τι μελέτε αντικτύπου που έχουν κάνει οι υπηρεσίε τη Κομισιόν. Να δούμε τι τροπολογίε που έχουν κάνει και άλλε επιτροπέ. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος νομίζω υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της όταν μιλεί για οικονομική ευθύνη και πρέπει να το παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό και η νομική επιτροπή ίσως και αυτή υπερβαίνει τα δικά της όρια αρμοδιότητας. Δεν υπάρχει ασφαλιστική αγορά για να ασφαλίσει τις, ε, τους κινδύνους αυτούς. Νομίζω, νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα η πρότυπα ασφαλείας με τρόπο που να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και να το καθιστά σχετικά εύκολο για τις χώρες που έχουν υψηλά πρότυπα ασφαλείας να τα τηρούν και βεβαίως να αρθούν σε υψηλότερα επίπεδα τα πρότυπα ασφαλείας όλων έτσι ώστε να μπορούν να εξορίζονται φυσικά αέρια και καύσιμα και σε άλλες περιοχές, άλλες θαλάσσιες περιοχές. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, Κύριε Αντρέας Μπαρέα σύντομα μόνο μερικά σχόλια. Και το λέει και στις τροπολογίες ο εισηγητής. Το θέμα της εταιρεία ε, τεχνική και οικονομική επάρκεια. Γιατί πολλές φορές γίνονται γεωτρήσεις διερευνητικές ε, που δεν είναι άρτιες από πλευράς τεχνικής, τεχνολογικής. Και ποιος φέρει την ευθύνη μετά όταν εγκαταλείπονται. Είναι και η τεχνική ευθύνη και η οικονομική και η αστική ευθύνη. Θα πρέπει όταν γίνεται μία γεώτρηση να υπάρχει βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό, θα είναι ε, επαρκές στο κοίτασμα για να είναι βιώσιμη εκμετάλλευσή του. Λοιπόν, από πλευράς περιβάλλοντος με ενδιαφέρουν αυτά και θα αναφερόμουν και στην τροπολογία 228 που αφορά το δίκτυο Natura. Γιατί υπάρχουν και διερευνητικές ε, ε, γεωτρήσεις, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τον τουρισμό, με το περιβάλλον ή μπορεί να υπάρχουν εργοστάσια αφαλάτωσης εκεί. Τι γίνεται αυτό. Και το θέμα του μείζωνος του μεγάλου ατυχήματος είναι επίσης πολύ σημαντικό. Γιατί όχι μόνο στη δική του χώρα και στη δική μου υπήρξε ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα οι ζημιές και παρακαλώ να προσέξετε την τροπολογία 228 και οι γεωτρήσεις, έστω και οι διερευνητικές, να ε, από εγγύσει από κάποια ασφάλεια. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ήθελα κάτι να ε, τονίσω, λέει ο κύριο Ανά. Μπορεί να έχουν γίνει πρόοδοι εδώ στην έκθεση, αλλά Τώρα ζητούμε υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας χωρίς να έχουμε πλειοψηφία στην Επιτροπή μας, έτσι ώστε οι ε, δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου να εντάσσονται στην νομοθεσία σε βέζο. Εάν θέλουμε αυτές οι δραστηριότητες να ε, πλαισιώνονται καλύτερα, εάν δεν θέλουμε η οικονομική εγγύηση να έρχεται εκ των να ενεργοποιείται γιατί πάντα είναι μετά το ατύχημα για τις αποζημιώσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε από πριν να έχουμε πολύ ψηλά πρότυπα ε, στη στιγμή της εκχώρησης, ε, ε, της παραχώρησης αυτών των δικαιωμάτων. Αλλιώς θα τρέχουμε να πληρώνουμε τα σπασμένα μετά. E Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας που πήραν μέρος στη συζήτηση και που έχουν καταθέσει τις τοπολογίες που έχουμε μπροστά μας. Κάποια σχόλια σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής και οι υπόλοιποι που πήραν μέρος από πλευράς Επιτροπής σας και κάποια θέματα τα οποία δεν τέθηκαν ίσως εκτενώς σήμερα, αλλά τα οποία ε, πρέπει να συζητηθούν για την επαλήθευση από ανεξάρτητους φορείς ή τρίτους φορείς. Πράγματι έχει μεγάλη σημασία η ανεξαρτησία εδώ της υπηρεσίας να ρυθμιστεί και νομοθετικά. Έχουμε εμπλακεί σε συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό με την ομάδα εργασίας για θέματα ενέργειας του Συμβουλίου. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε εμείς στην αρχή της ανεξαρτησίας. Είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να τεθεί από πλευρά της συγκεκριμένη νομοθεσίας που δεν λέγει στους, στις επιχειρήσεις το τι πρέπει να κάνουν αλλά ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους πρέπει να πετύχουν με τον πιο θα έλεγα ανεξάρτητο τρόπο με πιο αντικειμενικό τρόπο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των κινδύνων. Και μετά από αυτό να μην υπάρχει σύστημα, θα έλεγα, επαλήθευσης και από τις διάφορες υπηρεσίες και αρχές, έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαιτούμενες ή προαπαιτούμενες ανάγκες διασφάλισης της λειτουργίας για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Είμαστε υπέρ της ε, συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην διαδικασία, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης θαλασσίων περιοχών και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά και τους εργαζομένους της πλατφόρμες εξόριξης. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ήδη τμήματα νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπουν τη συμμετοχή των εργαζομένων και μεθοδολογία συμμετοχής τους στην ασφάλεια των μονάδων αυτών. Πρέπει να μην υπάρξουν επικαλύψεις με τις ρυθμίσεις αυτές και δεν θα πρέπει επίσης να υποβαθμίσουμε τα επίπεδα προστασίας που παρέχονται ήδη. Ίσως να υπάρχουν κάποια κενά, προσπαθήσαμε να τα καλύψουμε στην περίπτωση της συμμετοχής των εργαζομένων στην προετοιμασία της έκθεσης για τον λεγόμενο μίζονα κίνδυνο θέλουμε να βρούμε τι στοιχεία έχουμε στο κεντρικό θα έλεγα κόρπους των νομοθετικών μας για να προχωρήσουμε σε επιμέρους ρυθμίσεις. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην βλάψουμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την αρκτική ζώνη. Όλοι κατανοούμε βέβαια την ευαισθησία της περιοχής αυτής και είμαι και προσωπικά ε, υπέρ φυσικά του να υπάρξουν έλογες ρυθμίσεις για την περιοχή αυτή. Πιστεύω ότι η νομοθετική ρυθμίση όπως προτείνεται και η φιλοσοφία που υποβόσκει τη ρύθμιση αυτής θα πρέπει να καλύψει όλους τους τύπους του κινδύνου και τις ανάγκες όλων των ειδών του περιβάλλοντος στα πλαίσια των οποίων υπάρχει ε, δραστηριότητα επαγγελματική. Δεν υπάρχει εδώ μια απαρίθμηση των, του τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση, αλλά η υποχρέωση να αναλύσει όλες τις μορφές κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η προσφυγή σε ανεξάρτητες υπηρεσίες αξιολόγησης αν εξατληθούν όλες οι ίδιες δικές της δυνατότητες και σωστός εντοπισμός των κινδύνων. Και αυτό θα απαιτήσει, θα έλεγα, από πολλές επιχειρήσεις να αλλάξουν γενικά την οτροπία τους και να μπορέσουν να βρουν κανόνες λειτουργίας ακόμα και σε περιοχές πάρα πολύ σκληρές όπως τις γνωρίζουμε σήμερα ή σκληρές όπως θα τις γνωρίσουμε σε λίγο καιρό στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σε ζώνες όπως η Αρκτική. Για τους ορισμούς. Εδώ δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω ότι ό,τι είδαμε μέχρι τώρα στη Βόρεια Θάλασσα δεν θα καλυφθεί. Ο ορισμός που δίνουμε εμείς για το μείζον συμβάν λέμε ότι είναι το συμβάν το οποίο ε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην ίδια την μονάδα εξόριξης, στον έλεγχο της μονάδας εξόριξης ή προκαλεί διάχυση ε, προϊόντων ε, στο περιβάλλον. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει βέβαια να υπάρξει περισσότερη προσοχή σε σχέση με τους ορισμούς. Συναντώμεθα τακτικά με τα κράτη-μέλη και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας σε κάποια από τα θέματα τα οποία αφορούν τον ορισμό σαν παράδειγμα των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και εδώ είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Ένα θέμα το οποίο συνδέεται εν μέρη με το θέμα των ορισμών και δεν συζητήθηκε σήμερα τουλάχιστον επαρκώς ούτε σε επίπεδο ε, τροπολογιών είναι το θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών. Πώς ορίζουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσουμε ότι η έννοια των αρμοδίων αρχών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αν οι συνομοθέτες αποφασίσουν να προτιμήσουν την οδηγία γιατί τότε θα δοθούν περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη, οπότε οι αρμόδιες αρχές, αυτές που ονομάζουμε αρμόδιες αρχές, θα έχουν πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες και ο λόγος τους θα έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος. Θέλουμε λοιπόν αυτές οι ε, αρχές να είναι πλήρως ανεξάρτητες, να μην μπορεί να υφίστανται πιέσεις και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Τελευταίο θέμα, οδηγία ή κανονισμός. Είναι αλήθεια αυτά τα οποία ακούστηκαν από την κυρία Ριβάζη, ότι ένας από τους λόγους που προτείναμε τον κανονισμό είναι γιατί θεωρήσαμε ότι οι ρυθμίσεις οι νομοθετικές που φαίνεται ότι έρχονται στην επιφάνεια δεν παρέχουν πλήρως ε, ε, μια κάλυψη σχετικά με τους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να ισχύσουν. Απαιτείται λοιπόν ο κανονισμός. Η αδίποτε εναλλακτική πρόταση που να προτείνει την οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και ρυθμίσεις για το πώς θα βρούμε quick start λύσεις για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο άλλος λόγος που επιλέξαμε, για τον οποίο επιλέξαμε τον κανονισμό, είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε απευθεία σε επαφή με τη βιομηχανία, να νομοθετήσουμε με τρόπο άμεσα εφαρμόσιμο στις δραστηριότητες της βιομηχανικές, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση της οδηγίας τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες αυτές που παρέχει το κείμενο της οδηγίας, γιατί στόχος μας βασικά πρέπει να είναι η βιομηχανία και στον τομέα των δραστηριοτήτων σε θαλάσσιους χώρους. Ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν τέθηκε μέσω των τροπολογιών αλλά θα έρθει σε συζήτηση, είναι ο δυναμικός χαρακτήρας της νομοθεσίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, ιδιαίτερα αν επιλεγεί η οδηγία η νομοθεσία αυτή να είναι ανοιχτή προς το τέλος, δηλαδή να επιτρέπεται να εξελίσσεται με το χρόνο όσο εξελίσσονται οι τεχνολογίες, όσο οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για νέου τύπου δραστηριότητες αναπτύσσονται, εξελίσσονται και θα υπάρξουν και δευτερογενείς νομοθετικές εδώ ρυθμίσεις συμπληρωματικές της βασικής νομοθετικής ρύθμισης που συζητάμε τώρα. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα και για εφαρμαστικές συμφωνίες, όπως, αρμοδιότητες, όπως επίσης και για κατεξουσιοδότηση πράξης, οι οποίες θα σωρευθούν θα έλεγα και θα διευκολύνουν την λειτουργία της συγκεκριμένης οδηγίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητο πολύ περισσότερο στην περίπτωση της οδηγίας παρά στην περίπτωση του κανονισμού. Ευχαριστώ. Μπελέτ για να κλείσει η συζήτηση. Thanks, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάλυψω το πετάλεπτο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον κύριο Πανέκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα τελευταία σχόλια δηλαδή το δυναμικό χαρακτήρα και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Βεβαίως ε, το βλέπουμε αυτό με ανοιχτό πνεύμα, αλλά ίσως και η εντολή που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ευρεία. Πας θα βρούμε κάποια λύση. Σε ό,τι αφορά την αρμόδια αρχή και το σαφή ορισμό ε, και ιδιαίτερα την ανεξαρτησία των αρχών αυτών ε, στο πλαίσιο της οδηγίας. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο του όλου εγχειρήματο. Ε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες οι αρχές αυτές από οποιαδήποτε επιρροή ε, να εργάζονται εντός ενός πλησίου και θα πρέπει και η οδηγία αυτό να το προβλέπει. Συμφωνούμε πολύ με τα όσα λέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <coughs> Έχουν κάνει αντίστοιχε τροπολογίε και άλλοι συνάδελφοι και σίγουρα θα βρούμε κάποια ικανοποιητική λύση για τον ορισμό τη αρμόδια αρχή και το ρόλο που καλείται αυτή να διαδραματίσει. Τώρα οδηγία κανονισμό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι υπέρ ενός κανονισμού, ενώ στο Συμβούλιο είναι μάλλον ε, η συνένεση υπέρ της οδηγίας. Όχι. Συγγνώμη, διορθώνει ο μιλητής. Ναι, οδηγία έλεγα. Η συμμετοχή των εργαζομένων να μην υπάρχει επικάλυψη όντως και ε, να μην έχουμε νέα νομοθεσία που ανακαλύπτει κείμενη νομοθεσία ε, ε, ε, ίσως θα πρέπει να αφαιρεθούν αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα παραρτήματα και να μπουν στο διατακτικό για να καταλάβει και ο έξω κόσμος ότι πρόκειται για δέσμευση των ερετών εκπροσώπων για την ασφάλεια και τη συμμετοχή των εργαζομένων φυσικά. Τι ξέχασα. Α, η κυρία Φόρτ προτείνει πέρα από τη μελέτη αντικτύπου που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσουμε, λέει, εμείς, εδώ, από το Κοινοβούλιο, ξεχωριστή και ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών μελέτη αντικτύπου Και βέβαια, γιατί όχι, καλή πρόταση. Άλλο σημαντικό για τα πρότυπα των εταιριών που έχουν και παγκόσμιες δραστηριότητες, λεγόμενη παγκόσμια λοιπόν ευθύνη. Θα πρέπει αυτό να το ορίσουμε εμείς ότι ε, εταιρείε με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεούνται να τηρούν τα ίδια περιβαλλοντικά και αυστηρά πρότυπα ή απλώ να τι ενθαρρύνουμε. Γιατί δεν έχουμε την εξουσία να τι αναγκάσουμε. Ε, δεν έχουμε δηλαδή την, την, δικαιοδοσία. Ορισμένοι συνάδελφοι ε, θεωρούν ότι την έχουμε γιατί έχει γίνει και αλλού ε, αυτό. Παρακαλούμε λοιπόν την νομική υπηρεσία να ε, το ελέξει και να μας συμβουλεύσει σχετικά. Σίγουρα έχω ξεχάσει κάποια θέματα. Όπως σας είπαμε στην αρχή κυρία Πρόεδρε, Τη Δετάρτη συνεδριάζουν οι σκιώδεις και θα Είμαστε στη διάθεσή σας, ελπίζω να είναι επικοδομητική η συζήτηση, αλλά γενικά το πνεύμα που επικρατεί είναι θετικό για αυτή τη νομική πρόταση και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πριν την 9η Οκτωβρίου που θα έχουμε εδώ την ψηφοφορία όπως έχει προγραμματιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπελέτ. Όπως εσείς ο ίδιο υπενθυμίσατε η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή προβλέπεται την 3η 9 Οκτωβρίου. Τελειώσαμε το πρώτο τμήμα των εργασιών μας, θα ξεκινήσουμε σύντομα τις ψηφοφορίες. Θα πρέπει να περιμένουμε τρία λεπτά γιατί οι ψηφοφορίες προβλέπονται για την 16η απογευματινή ακριβώς. Θα δώσουμε τη δυνατότητα λοιπόν σε όλους όσους το επιθυμούν να έλθουν και θα κλείσουμε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. On a quatre Combien Dans la que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 Bene, allora possiamo iniziare il voto. Facciamo... Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ να υπάρξει έλεγχο των παρουσιών των πολιτικών ομάδων πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά τώρα λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Τριάντα δύο ψήφισαν. Ξεκινάμε. Eh, Η πρώτη ψηφοφορία σήμερα δεν είναι παρόν ο κ. Γιούκ. Χάουγκ, η κυρία Χάουγκ εννοεί η πρόεδρο, αλλά έχει αντικατασταθεί από την κυρία Καστίγιο. Α, ναι. Πρόκειται για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 81. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 82. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 84. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει γίνει δεκτή αλλά υπάρξει παρακαλώ μια ψηφοφορία ηλεκτρονική για την 85. Πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ 27 κατά. Απορρίπτεται η 85. 86 και 87 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 88. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 89 και 90 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Τροπολογία 91 και 92 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Τροπολογία 93 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 95 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 95. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 20 κατά. Συνεπώς γίνεται δεκτή. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98-99 από κοινού. Υπέρ. Α, μόνο την 98 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Την 100 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 8 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 101 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 9 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά 106 ψηφίστηκε η 107 τώρα 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 111 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 22 κατά. Ζητώ συγγνώμη, Ίσως λίγο με δικαιολογείτε βλέποντας τους αριθμούς αυτούς. Λοιπόν, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 124 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 125 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 128 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή 130 υπέρ κατά αποχές δεκτή 131 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές αδεκτή 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απδεκτή αλλά ας υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 155 πέραση ψηφοφορίας 26 υπέρ, 22 κατά δεκτή. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 158 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 159 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 160 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ για την 166 ηλεκτρονικός έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 20 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 και 69 μαζί ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή 172 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για το 172 21 υπέρ 27 κατά περίφθη, 173 υπέρ κατά αποχές δεκτή, απορρίπτεται συγγνώμη, 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 176 και 77 μαζί υπέρ κατά αποχές αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα της ψηφοφορίας. 35 υπέρ 13 κατά δεκτή. 178 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 179 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 181 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση ψηφοφορία 7 υπέρ 41 κατά. Συγγνώμη συνάδελφοι, αλλά δεν ψηφίσατε γρήγορα. Λοιπόν, απερίφθη 181, περνάμε στην 182, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 184, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 και 86 μαζί υπέρ κατά αποχές απερίπτεται δεκτές 188 τώρα α όχι γυρνάμε πίσω στην 185-186 από κοινού ξεκινάμε Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 20 κατά. Δεκτές. Περνάμε στην 188 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. 189. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 190. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 191. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 193 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 195 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 196 υπέρ κατά αποχές απερίπτεται, 197 υπέρ κατά αποχές δεκτή 198 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 199 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 200 υπέρ κατά αποχές δεκτή 201 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 202-203 μαζί ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 204 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 205 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 206 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 207 υπέρ και 8 μαζί κατά αποχές δεκτές 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή 211 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 212 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 213 με μία προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 215 υπέρ κατά αποχές απερίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απε, δεκτή 14 υπέρ κατά δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 216-17 και 218 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 219 υπέρ κατά αποχές δεκτή 220 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 221 υπέρ κατά αποχές δεκτή 222 υπέρ κατά αποχές δεκτή 223 υπέρ κατά αποχές δεκτή 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 226 υπέρ κατά <coughs> αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 227 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2.29 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 219 τώρα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 231 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 232 υπέρ κατά αποχές δεκτή 233 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 234 υπέρ α όχι η 34 δεν ψηφίζεται η 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 237 υπέρ κατά αποχές δεκτή 238 υπέρ κατά αποχές δεκτή 239 υπέρ κατά αποχές δεκτή 240 υπέρ κατά αποχές δεκτή θα πρέπει να συγγνώμη ξέχασα σε αυτή τη σελίδα να ψηφίσουμε το 2.34 παρακαλώ, πρέπει να την ψηφίσουμε 2.34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αλλά πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Κιούζα 23-24 υπέρ 24 κατά περίφθη με μία ψήφο. Περνάμε τώρα στο 2.41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.45 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 2.46 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 2.46 υπέρ, κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34, 35 μάλλον υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 ε, μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την 36. Ελέγχουμε την 36. Votazione chiusa. Πέρα της ψηφοφορίας, 33 υπέρ, 15 κατά γίνεται δεκτή 36. Ψηφίσαμε την 35, ακούγεται μια ερώτηση. Ψηφίσαμε μόλις τώρα την 36, λέει η κυρία Σαρτόρη. Την 35 την είχαμε ψηφίσει πριν, τώρα την 36. 37 λοιπόν τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν απερίφθη. Τροπολογία 39. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 44. Υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 45. Υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 46. Υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 47, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Κοιτάξτε, εσείς ζητήσατε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 47. 4, 7, 47. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία λέει η Πρόεδρος. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία γιατί υπήρξε μια κάποια σύγχυση. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την τροπολογία 47. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 36 υπέρ 11 κατά δεκτή. Καλώς λοιπόν συνεχίζουμε με την 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τοπολογία. 1 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ εναντίον αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 51 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 52 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 53 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 54 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 55 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται 3 με μια προφορική τροπολογία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 4 ε, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73-74 υπέρ Α, όχι, μόνο την 73, έκανα λάθος. Μόνο η 73 ψηφίζεται. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή όχι ηλεκτρονικός έλεγχος για την 76 παρακαλώ 76 ελέγχουμε τέλος της ψηφοφορίας 40 ή κατά 8 υπέρ απερίφθη. Λοιπόν, τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψήφος. Άρχεται ψηφοφορία. καλός. Πέρα της ψηφοφορίας. 40 υπέρ 6 κατά 2 αποχές έγινε δεκτή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της εκθέσεως Μπαλτσίτης. Δεν ξέρω αν έχετε τον κατάλογο όλοι. Έχουμε την έκθεση Μπαλτσίτης, τροπολογία 30, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 31 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 34 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 35 υπέρ, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34 βέβαια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 28 υπέρ 19 κατά. Η 34 γίνεται δεκτή. Η τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά δεν ελέγχω απόλυτα. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 37. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ 26 κατά περίφθη. Τριάντα οκτώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 in tre parti. Prima parte, a favore. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, <clears throat> α μια στιγμή. Κοιτάξτε πρέπει να ψηφίσουμε την 40. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ, <clears throat> κατά, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 τώρα, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45, 49 μάλλον υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 51 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 52 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές αποχές επαναλαμβάνω δεκτή. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 83. πέρα της ψηφοφορίας 29 υπέρ 18 κατά. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά δεκτή. 3 υπέρ κατά δεκτή. 21 υπέρ κατά δεκτή. 4 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά δεκτή. 3 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά δεκτή. 6 υπέρ κατά δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Λοιπόν, 40 υπέρ 6 ε, κατά 2 αποχές. Η τρίτη ψηφοφορία είναι η ψηφοφορία Έντι Τέρτσοκ. για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως για την 2. Τέλος της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ συγγνώμη την 8 ψηφίζουμε ψηφίζουμε την 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε τώρα στην 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές δε, απορρίπτεται. 14 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 παρακαλώ. 26 26 υπέρ 22 κατά. 23. 23 λοιπόν. Α, έκανα λάθος λέει. Πρόεδρος το 24, 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 25. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 26, 27 μάλλον υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Μετά από την 27 πηγαίνουμε στην 32. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 26 λέει η πρόεδρος. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την 28 όμως. Επανέρχεται 28 υπέρ. Όχι. Λάθος λέει η πρόεδρος. Σταματάει, ζητάει χρόνο. 32. 32 il faut voter, Le 32. 32. Le 32. Allora, passiamo al 32. Περνάμε στην 32. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 35, υπέρ, κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία α κάποιος έχει στο το λόγο Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια θέλω να κάνω δήλωση ότι τούτη εδώ η Επιτροπή φαίνεται ότι συμφωνεί αν θέλουμε να είμαστε υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων θα πρέπει να έχουμε το ίδιο μήνυμα και το Συμβούλιο. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουμε όλα τα χρήματα για την έρευνα, για τη ε, διασύνδεση ε, ε, της Ευρώπης, για όλη την έρευνα. Αυτό ψηφίζουμε και με την τελική ψηφοφορία αυτό διατρανώνουμε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία τελική. Τέλος της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, 4 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Και τώρα περνάμε Στην ψηφοφορία του συνάδελφη Beauty Coffer, μία ψήφος μόνο, τελική ψήφος, ηλεκτρονική ψήφος για την έκθεση Beauty Coffer. Τέλος της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την προσοχή τους. Περνάμε λοιπόν τώρα. Στη συνάδελφο Τζόρνταν. Αλλά ας περιμένουμε ένα λεπτό γιατί κάποιοι θέλουν να φύγουν. Per quelli che devono abbandonare l'aula prima di iniziare. Minuto. Η πρόεδρο, τώρα τον λόγο έχει η κυρία Τζόρνταν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον Αύγουστο, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τον οργανισμό ΆΣΕΡ, Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Πρώτη επίσκεψη αυτή σε ένα οργανισμό που ήδη ε, λειτουργεί εδώ και ένα έτος περίπου στη Λιουμπιάνα. Η αντιπροσωπεία ήταν εγώ, Σμιθ, Ντουρρόνικ από την Γραμματεία και Σπίλερ Μάιζεν και ένας βουλευτής ακόμη. Συναντηθήκαμε με τον Αλμπέρτο Ποτότσνικ που είναι πρόεδρος της Acer ή του Acer και τον πρόεδρο του Board of Regulators, καθώς επίσης τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριο Βόσνιακ. Στη διάρκεια της επισκέψεως μας συνόδευε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς ε, συνομιλήσαμε μαζί τους για εφαρμογή αρχών της ενιαίας αγοράς Μιλήσαμε λοιπόν για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στο ηλεκτρικό ρεύμα και, και στο φυσικό αέριο, για τα σχέδια ανάπτυξης των ενεργειακών συστημάτων, για τις σχέσεις μεταξύ του Acer και των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ σύντομα, λίγα λόγια για τις συνομιλίες αυτές. Πρώτα, η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πολιτικός στόχος ότι δηλαδή η ενιαία αγορά να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2014. Ο διευθυντής Ποτότσνικ ανέπτυξε με λεπτομέρεια τις δραστηριότητες του οργανισμού τους που συντάσσουν πλαίσια για τα δίκτυα αυτά. Αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές θα αποτελέσουν την βάση επί της οποίας θα οικοδομήσει ο Acer τα σχέδια για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο και μετά θα περάσουν βέβαια από τη διαδικασία επιτροπολογίας. Ο Acer στο τέλος θα γνωμοδοτήσει. Για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζονται οι συνομιλίες, η εργασία προχωρεί ομαλά και εκτιμάται ότι μέχρι το 2013 θα έχει ολοκληρωθεί. Στον τομέα του φυσικού αερίου η διαδικασία είναι ωστόσο πολύ πιο αργή. Μόλις φέτος στο φόρουμ της Μαδρίτης λήφθηκε η απόφαση να συνταχθεί ένας οδικός χάρτης. Ωστόσο το έργο καθυστερεί. Άλλος τομέας που μας απασχόλησε στις συνομιλίες αυτές ήταν η εφαρμογή του REMIT, του κανονισμού δηλαδή, που θα πρέπει να εφαρμοστεί και όταν θα εφαρμοστεί θα αποτρέπει τις καταχρήσεις στην αγορά και τις περιπτώσεις απάτης. Βέβαια αυτό θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση. Σύμφωνα με τον οργανισμό Acer, πρόκειται από τις πιο σημαντικές προκλήσεις τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Και αναμένουν ότι καθημερινά θα ελέγχουν περίπου 500.000 συναλλαγές το σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτουν υποτίθεται ότι θα το κάνει αυτό συν 100.000 συναλλαγές καθημερινά που θα τις επεξεργάζονται άνθρωποι. Γι' αυτό η εφαρμογή του Remit είναι πολύ σημαντική υπόθεση και προϋποθέτει την αγορά ε, υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και λογισμικού και βέβαια πρόσληψη επαρκούς προσωπικού. Βέβαια ο προϋπολογισμός που προβλέπεται είναι περιορισμένος και υπερβολικά χαμηλός για να ανταποκριθεί ο οργανισμός σε όλες αυτές τις ε, ανάγκες. Εμείς εγκρίναμε έναν προϋπολογισμό υψηλότερο κατά 3 εκατομμύρια ευρώ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και τους συναδέλφους μας της Επιτροπής Προϋπολογισμών ώστε να εγκρίνουν το ποσό αυτό και να αποφευθεί έτσι οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αγορά τεχνικών υπολογιστών και λογισμικού. Βέβαια, το θέμα του προσωπικού θα παραμείνει διότι θεωρούν ότι χρειάζονται 50 ε, υπαλλήλους για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Ωστόσο, το, η τεκμηρίωση, η σχετική μάλλον ε, νομοθεσία, η, ο, οι κανονισμοί που υπάρχουν για την, για την ώρα, ε, προβλέπουν μόνο 15 θέσεις. Τώρα, ο οργανισμός για τη σχετική υποδομή έχει κληθεί να συντάξει γνωμοδότηση και αυτή είναι σημαντική πρόκληση. Και η σημαντική αυτή πρόκληση έγκυται στο πώς θα εξασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των έργων, των project που έχει αναλάβει με ταυτόχρονα ανάπτυξη επαρκούς μεθοδολογίας η οποία να διασφαλίσει την ε, τελική επιλογή και αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών. Επίσης, η ένταξη των διαφόρων εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα, σύστημα ενέργεια, στα συστήματα διανομής ενέργειας και αυτά βέβαια είναι γνωστές προκλήσεις και έχουν σχέση με την ανάπτυξη των δικτύων που θα εξασφαλίσουν επαρκή ικανότητα επαρκή, capacity δηλαδή στην αγορά. Θα πω λίγα για το ιδιαίτερο αυτό θέμα στο τέλος της παρεμβάσεώς μου. Επίσης, υπάρχει και η συνεργασία του Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών με τον Acer. Η συνεργασία αυτή είπαν ότι είναι καλή. Η συνεργασία με τους εθνικούς συντονιστές είναι καλή. Επίσης, το Συμβούλιο αυτό αποτελείται από 29 ευρωπαϊκές χώρες, περισσότερες από τις 27. Οι εθνικοί ρυθμιστές αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με του Acer. Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης βέβαια το έργο τους έχει πολλαπλασιαστεί. Αντιμετωπίζουν όμως και μεγάλες δυσκολίες ό,τι αφορά την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Μιλήσαμε και για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Acer, που μέχρι τώρα η συνεργασία αυτή ήταν καλή και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει με τον τρόπο αυτό να χρησιμοποιήσει ακόμα, να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Μιλήσαμε και με όλους τους υπαλλήλους του Acer, είχαν προσκληθεί όλοι να μας συναντήσουν. Συναντηθήκαμε μαζί τους στη μεγαλύτερη αίθουσα που διαθέτουν και ήρθαν σχεδόν όλοι. Εγώ εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τον ζήλο τους, γιατί τα πρόσωπα αυτά πραγματικά ε, έχουν τη διάθεση να δουλέψουν σωστά. Θα τελειώσω λέγοντας ή μάλλον αναφέροντας ορισμένες συστάσεις προς την Επιτροπή μας. Ε, συστάσεις που ελπίζω ότι θα συζητηθούν και στην συνάντηση των συντονιστών. Στο τέλος δηλαδή των συναντήσεών μας υιοθετήθηκαν ορισμένα συμπεράσματα. Είπαμε ότι επιθυμούμε οι επαφές μεταξύ της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ήτρε, συνεργασίας δηλαδή με τον Acer και ε, από την άλλη μεριά με τον Acer, να γίνουν πιο ζωντανές, πιο ζωηρές είπαμε να κάνουμε δύο ή τρεις συναντήσεις. Εν τέλει συμφωνήσαμε ότι θα προτείνουμε να συναντώμαστε, να δύο φορές τον χρόνο και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Ο ACER, ο Οργανισμός ε, δηλαδή Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ενέργειας θα μας εξηγεί πώς κατά την άποψή του θα, ποιες μάλλον θα είναι οι επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας. Προτάθηκε επίσης να συναντώμεθα συχνότερα με τους εκπροσώπους του ε, Διοικητικού Συμβουλίου. Και μια τρίτη πρόταση που έγινε ήταν η Επιτροπή Ήτρε να χρησιμοποιήσει καλύτερα την τεχνογνωσία του οργανισμού. Δηλαδή να του ζητούμε γνωμοδοτήσεις. Είπαν ότι πολύ ευχαρίστως θα μας ε, δίνουν τις γνωμοδοτήσεις τους. Επίσης, ε, κάναμε και συνέντευξη τύπου στο τέλος της επισκέψεως και με την ευκαιρία θα προτείνω τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συντάσσουν πάντοτε ή μάλλον να διοργανώνουν πάντοτε ε, συνέντευξη τύπου όταν μια αντιπροσωπεία της Ήτρε επισκέπτεται μια χώρα. Κάτι που νομίζω ότι δεν έχει γίνει πάντοτε μέχρι τώρα. Ωστόσο το, το συνιστώ πολύ θερμά διότι η ανταπόκριση των δημοσιογράφων ήταν πολύ ε, έντονη. Και θα ευχαριστήσω βεβαίως όλες και όλους όσοι συμμετέσχουν στην ε, αντιπροσωπή αυτή, καθώς επίσης και τα μέλη της γραμματείας που μας συνέδραμαν σημαντικά. Εσείς κύριε Τούρμες. Πρώτα θα πω ότι η αντιπροσωπεία ήταν μεν μικρή, αλλά η δράση της αποτελεσματική και με μεγάλη με ευχαρίστηση πήγα μαζί με την κυρία Τζόρνταν ε, στην ιδιαίτερη πατρίδα της που αυτό ήταν ένα ε, συν νομίζω ότι δουλέψαμε σκληρά αλλά ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα η έκθεση τα λέει λίγο πολύ όλα αυτό που θέλω να πω εγώ είναι και να τονίσω είναι ότι ο οργανισμός Acer παίζει τόσο κεντρικό ρόλο για την μεταφορά στα εθνικά δίκαια των ε, δεσμών ε, ε, ρυθμίσεων και κυρίως για τα διοικητικά. Γιατί για μας το πρόβλημα, με εμάς που είμαστε policy makers, είναι ότι αν δεν μας εξηγήσουν καλά, τα χάνουμε λίγο, χανόμαστε. Συχνά τα πράγματα φαίνονται πρώτης όψεως τεχνικά αλλά εδώ μιλούμε για μια αγορά αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα λοιπόν όσα κρύβονται πίσω από τεχνικά επιχειρήματα πολύ συχνά είναι και πολύ πολιτικά. Γι' αυτό μπορούμε να ζητούμε τη γνωμοδότηση του Acer και να του ζητούμε να μας υποβάλουν σύντομες συνόψεις που να εξηγούν και ποια είναι τα πολιτικά καυτά θέματα που κρύβονται πίσω από κάποιους κώδικες. Γιατί αλλιώς για μας είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει. Ένα σημαντικό θέμα είναι βέβαια η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του REMIT. Ως συνομοθέτες έχουμε αναλάβει τεράστια ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετούμε και μετά να μην βρίσκουμε ούτε 5-6 εκατομμύρια ευρώ το πολύ για να χρηματοδοτήσουμε την απαραίτητη ε, επένδυση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μηχανογραφικά συστήματα και στα πρόσωπα τα οποία είναι απαραίτητα. Εάν σε δύο ή τρία χρόνια κάποιος ανακαλύψει μια μεγάλη απάτη στα ευρωπαϊκά συστήματα διανομής ενέργειας. Θα δακτυλοδεικτούμε τότε τους Υπουργούς Οικονομικών οι οποίοι δεν επέτρεψαν να μπουν στον προϋπολογισμό του 2013 τα 5 ή 6 εκατομμύρια που ήταν απαραίτητα για την εφαρμογή του REMIT. Δεν είναι δυνατόν κυβερνήσεις να συνομοθετούν μαζί μας για την ορθή εποπτεία της αγοράς ενέργειας και μετά να περικόπτουν τα κονδύλια τα 5-6 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του κανονισμού REMIT. Οι αιτήσει εκθέσει του Acer για φέτο ήταν καλά, διότι ήρθαν εδώ και μα τα υπέβαλαν. Νομίζω ότι ήρθαν όμω περί τα τέλη του Ιουνίου, έκτου δηλαδή, που είναι δύσκολη στιγμή για μας. Α του γράψουμε ένα γράμμα, και εσείς η Προεδρία δηλαδή, στο όνομα της Επιτροπής μας, ότι καλή ήταν η συνδρομή τους του περασμένου έτους, αλλά προτιμούμε να είναι περί τα τέλη Μαΐου, γιατί αλλιώ για μας είναι δύσκολο να οργανωθούμε έγκαιρα ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Και επίσης η κυρία Τζόρνταν τόνισε ότι έχουμε και δουλειά να κάνουμε. Και δείχνω εδώ τον Giles Τσίτσεστερ που είναι συντονιστής της ομάδας επαφής με τον Acer εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε δύο-τρει συναντήσεις τον χρόνο και η τελευταία θα πρέπει ε, να αφιερώνεται και στην έκθεση για τον επόμενο χρόνο, όπως είπα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και να λύσουμε το πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε λύσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχουμε δύο εκπροσώπους που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Acer. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να έρθουν στην ομάδα επαφής Acer διότι το κοινοβούλιο δεν τους έχει, δεν έχει προβλέψει τον απαραίτητο μικρό περιπολογισμό για να πληρώσει το ταξίδι τους στις Βρυξέλλες. Στην ομάδα επαφών με τον Acer ε, τουλάχιστον αυτή η ομάδα επαφών πρέπει να μπορεί να συζητήσει με ορισμένα πρόσωπα για το ποιε θέσει προβάλλουν εκπροσωπώντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουμε εμεί ποιε είναι οι θέσει του και δεν γνωρίζουν αυτοί απαραίτητα ποια είναι η δική μα θέση. Να λοιπόν κάτι επί του οποίου πρέπει να επανέλθουμε στο επίπεδο των συντονιστών. δεν φταίνε οι συντονιστέ τη Ήτρε, ούτε η γραμματεία που δεν βρήκαν λύση, αλλά οι διοίκηση του Κοινοβουλίου σε υψηλότερο επίπεδο. Χρειαζόμαστε όμω μια λύση. Αλλιώ δεν έχουμε επαρκή επαφή μεταξύ των εκπροσώπων μα. Interface στα αγγλικά. Ε, νομίζω ότι μπορώ να αρκεστώ σε αυτά τα λόγια. Ε, ναι. Ο κύριος Τσίτσεστερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την κυρία Τζόρνταν για την ε, παρουσίασή της και ε, για την εξαιρετική επίσκεψη ε, στο ΙΣΕΡ. Θα ήθελα και εγώ να είχα πάει, αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις και όλα. Πολύ καλό λοιπόν που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε σύντομα να πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, υποστηρίζω πλήρως τα επιχειρήματα που ακούσαμε και από τη Ρωμάνα και από τον Κλοντ σχετικά με τη λειτουργία του REMIT στον είσαι. Πώς να το πω. Οι νομοθέτες έχουν μια κακιά συνήθεια. Φορτώνουν τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες με απαιτήσει χωρίς να τους δίνουν τους απαραίτητους πόρους για να ανταπεξέλθουν. στην περίπτωση αυτή, το τόνισε και ο Κλοντ Τούρμες, ότι χρειάζονται επιπλέον πόρους, που δεν είναι και πολλά τα χρήματα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη λειτουργία της παρακολούθησης και του ελέγχου της αγοράς. Οπότε θα παρακαλούσα και εγώ να υπάρξει μια τέτοια πρόβλεψη στον προπολογισμό. Αυτό ήταν το πρώτο μου. Δεύτερο, θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω και ευχαριστώ τον Κλώτ που μου το θύμισε ότι είμαι πρόεδρος της εν λόγω εργασίας για το πόσο ε, σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την επαφή μας ε, από την Επιτροπή εδώ με τον ΕΙΣΕ. Όταν ε, κάναμε την ομοθεσία και εγώ ήμουν τότε εισηγητής, είχαμε συμπεριλάβει αρκετές διατάξεις για να τους δίνουμε την ευκαιρία μας χρησιμοποιούν εμάς ως ένα όργανο αναφοράς για να υπάρχει μια απόσταση ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να τους ε, ενισχύσουμε, να τους ενθαρρύνουμε και να τους παροτρύνουμε να έρχονται ε, να ε, τα συζητούμε. Εγώ θα προτιμούσα τρεις φορές το χρόνο, έστω και δύο, εντάξει, αρκεί. Αλλά να δούμε πότε θα πρέπει να διεξάγονται. Γιατί αγωνιζόμαστε κάθε φορά και φέτος να βρούμε το σωστό χρόνο. Φαίνεται καθυστερήσαμε φέτος. Ίσως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με τη γραμματεία για το 2013. Και ένα τρίτο που μου θύμισε ο Κλοντ. Το θέμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Είχα μεγάλη δυσκολία σε σχέση με τις ταξιδιωτικές δαπάνες των δικών μας ε, υποψηφίων και δύο από τους προηγουμένους που είχαμε διορίσει, που είχαμε προτείνει, ανήθηκαν γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι με την αποζημίωση που ε, θα έπαιρναν για τα ταξιδιωτικά τους έξοδα. Και ε, δυστυχώ υπάρχει ο περιορισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποια έξοδα επιστρέφονται, αποζημιώνονται και καλύπτονται. Λυπάμαι λοιπόν, λοιπόν που παραμένει αυτή η κατάσταση. Ε, ψάξαμε και δυσκολευτήκαμε πολύ να το λύσουμε. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα πρώην τμήματάρχη μας, τον κύριο Λοή Ματινουά, ε, που νομίζω ζει στις Βρυξέλλες, οπότε θα μπορούσε να συμμετέχει ε, στη συνεδράση της Επιτροπής μας και καλό θα ήταν να τον καλέσουμε να μας πει πώς βλέπει εκείνος ε, τη λειτουργία του οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνάντηση των συντονιστών θα τεθεί το θέμα. Η κυρία Χέρτσοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Για πολύ καιρό ε, δεν ασχολήθηκα με θέματα δημοσιονομικά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, γιατί ήμουν αρμόδια για θέματα βιομηχανίας. Αλλά τελικά έμαθα ότι όλα τα θέματα για να λειτουργήσουν θέλουν τον προπολογισμό τους. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον Acer. Ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός, έγινε μεγάλη συζήτηση νομοθετική και υποσχεθήκαμε στον Ευρωπαίο πολίτη ότι είμαστε υπέρ της διασυνοριακής αγοράς ενέργειας. Και την προηγούμενη θητεία όσοι ήσασταν εδώ θα θυμάστε τι περίφημη αρχή για το πώς ήταν δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να βρεθεί ο σωστός οργανισμός. Και ρωτώ, πώς φανταζόμαστε ε, την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη να λειτουργήσει αν δεν έχουμε λίγα εκατομμύρια για μια διασυνοριακή ε, λειτουργία, ένα οργανισμό που τα διαχειρίζεται αυτά που λέγεται ίσε. Λοιπόν, όταν νομοθετούμε θα πρέπει να συνοδεύεται αυτό από τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Και για τον προπολογισμό του 2013 που μόλις ψηφίσαμε ε, με τον κύριο Πιτικόφερ και τη δική μου έκθεση. Τι θα γίνει αν δεν τα συζητούμε αυτά σε βάθος, αλλά είμαστε επιπόλαιοι. Προτείνω όλες οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουμε ένα σχέδιο τροπολογίας για τον προπολογισμό και να μην αφήσουμε μόνο του τον ε, αρμόδιο εισηγητή για θέματα οργανισμών να υπερασπιστεί τον ΕΙΣΕ. Παρακαλώ να συνυπογράψουμε την τροπολογία αυτή στον προπολογισμό και να στείλουμε επιστολή για να δείξουμε στον κόσμο ότι το επιδιώκουμε. Και να μάθουμε και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί σήμερα γίνονται πολλές απόπειρε από το κεφάλαιο 1α να φύγουν χρήματα, μάλλον να καλυφθούν από το κεφάλαιο 5 από την κατηγορία 5, αλλά αν μειωθεί εκεί το ανθρώπινο δυναμικό δεν θα μπορούμε να υλοποιούμε σωστά τις πολιτικές. Χρειάζεται λοιπόν να συμφωνήσουμε καταρχήν και να υλοποιούμε σωστά και να εφαρμόζουμε την νομοθεσία και δεν ε, υποχωρούμε ούτε συμβιβαζόμαστε για θέματα προπολογισμού. Και ζητώ συγγνώμη από το Συμβούλιο, το ξέρω ότι και αυτοί τα λεφτά τους σκέφτονται, αλλά δεν γίνεται. Πώς θα εφαρμόσουμε τις πολιτικές που αποφασίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι για όλους είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει πλήρως ο οργανισμός Acer και με σωστό τρόπο. Και γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε με την απόσπαση των δικών μας στο Συμβούλιο το διοικητικό είχαμε δύο ευρωβουλευτές που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και τελικά υποχρεώθηκαν να καταθέσουν την εντολή τους και να αρνηθούν τη συμμετοχή, οπότε δεν συμμετέχει καθόλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια διορίστηκε κάποιος αντικαταστάτης με ε, την υπόσχεση ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο στάθηκαν ικανοί να κάνουν μέχρι σήμερα αυτή τη βελτίωση, ούτε να την επιβάλλουν. Γιατί είναι και θέμα αρχής. Ένα δεύτερο τώρα. Ο οργανισμός ACER ε, θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκός οργανισμός, οπότε ε, και τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν να συμμετέχουν, δεν ξέρουμε ποια μορφή, αυτό το καιρό γίνονται διαπραγματεύσει για μεγάλη ενεργειακή συμφωνία, ιδιαίτερα με την Ελβετία, όπου προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο επίτροπο Τιγκέρ να ε, ε, μην το θεωρήσει αμυγός ε, ενεργειακή πολιτική, αλλά μια σημαντική πρόοδο στις σχέσεις με την Ελβετία, ιδιαίτερα στις διαδικασίες διακανονισμού των διαφόρων. Βέβαια, εδώ ε, από αυτό το στοιχείο περιπλέκονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά ελπίζω ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος να ειδωθεί συνολικά και να συμπεριληφθεί αντίστοιχα ε, στον Acer και η Ελβετία. Νομίζω θα ήταν κάτι ευπρόσδεκτο αυτό για όλους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα. Θα ήθελα μόνο να υποστηρίξω θερμά την πρόταση της κυρίας Χέρτσοκ. Ο κύριος Τούρμες στα γερμανικά. Άκουσε κύριε Ρούμπικ βέβαια να συμμετάσχει κάποτε η Ελβετία στον Acer όχι να εκμεταλλεύεται μόνο τις θετικές πλευρές, αλλά πρώτα χρειαζόμαστε τη συμφωνία με την Ελβετία και μετά να έρθουν στον Acer. Αλλιώς, ε, εάν μπορούν να συμμετάσχουν στα πάντα, χωρίς πρώτα να υπογράψουν τη συμφωνία, και αν δεν υπογράψουν ποτέ, διότι υπάρχουν δυνάμεις στην Ελβετία που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία για την ενέργεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσέξουμε λοιπόν να μην τους δώσουμε όλα όσα θέλουν πριν υπογράψουν τη συμφωνία. Τέλειωσε λοιπόν η συζήτηση εδώ. Ευχαριστούμε τους ε, συμμετασχόντες. Ο κ. ποτέ είναι εδώ, θέλει να, να μιλήσει. Όχι. Καλά. Τον ευχαριστούμε και κλείνουμε εδώ την ενημέρωση για την επίσκεψη στον Acer. Και το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης είναι... Η κυρία Τεκαστήγιο Abbiamo il rendiconto della delegazione della Commissione ITRE a Riga. Για την αποστολή της ΙΤΕ στη Ρίγα, η κυρία Δεκαστήγιο δεν είναι ανάμεσά μας. Η Αντευσδοτήρ, θέλετε κάτι να πείτε. Έχουμε στείλει νομίζω γραπτή ενημέρωση για την αντιπροσωπεία μας εγώ, η κυρία Τροτμάν, πήγαμε και η κυρία Πιλάρ Δελ Καστίγιο. Συναντηθήκαμε με ε, εκείνους που μας είπαν ε, πώς λειτουργεί ε, και είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα με το άρθρο 7 και την αντίστοιχη διαδικασία και τόνισαν ότι είναι πολύ προβληματική. Αλλά γενικά δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Είδαμε και τη ρυθμιστική αρχή της Λετωνίας για τις τηλεπικοινωνίες και μας ε, ε, είπαν για το κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα ότι θα πρέπει να ε, δούμε κάποια θέματα απάτης για τον τερματισμό της λειτουργίας. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και κατά με τον Πρωθυπουργό της χώρας που μας είπε και αυτό διαφορετικά και γενικά δεν νομίζω ότι ήταν η επίσκεψη πολιτικά έτσι πάρα πολύ επίμαχη με κανένα τρόπο. Νομίζω ότι, ότι τις ρυθμίσεις ευνοούνται περισσότερο κάποιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με κάποιες άλλες για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αποστολής. Καλώς. Ευχαριστώ. Έπρεπε να φύγει η κυρία Δεκαστήγιο, αλλά μου είπε ότι όλοι οι συναδέλφοι, σε όλους τους συναδέλφους μάλλον, έχει αποσταλεί ένα σημείωμα, οπότε τελειώσαμε πλέον τις εργασίες μας. Η επόμενη συνάντησή μας είναι την 8η Οκτωβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 για να συνεχίσουμε. Για Συνεχίζετε και την 9η βέβαια.